Σας ε, καλωσορίζω στην τελευταία συνεδρίαση της ΠΕΤΗ πριν από τις καλοκαιρινές δικοπές. Σας είμαστε έτσι ευχάριστοι και χαλαροί εν ώψη και των ε, διακοπών που έρχονται. Πρώτα απ' όλα όμως θα ολοκληρώσουμε την ημέρα διάταξη σήμερα. Θα συναντήσουμε πολύ ενδιαφέροντες ε, αναφέροντες. Και εδώ, α, μου φέρανε και σφυράκι. Αρχικά, σημείο 2, υιοθέτηση της μέσης διάταξης. Ας περάσουμε στο, να, μάλλον, να μεταφέρουμε τα σημεία 5 και 6 για σήμερα το απόγευμα, για πρακτικούς λόγους, ακριβώς πριν την ψηφοφορία για την απόφαση ψηφίσματος ε, και προφορικού ερωτήματος. Καλύτερα είναι να συγκεντρώσουμε μαζί τις ψηφοφορίες μια και έξω για να μην ε, αναγκάζουμε του συναδέλφου να πηγαίνουν έρχονται συνεχώ. Αν συμφωνείτε κι εσεί, ε, ωραία, ευχαριστώ. Μετά να κρίνουμε τα πρακτικά τη συνάντηση του Μαΐου και του Ιουνίου, σημείο 3. Τα έχετε δει. Τα πρακτικά έχουν ε, μοιραστεί και για το Μάιο Υπάρχει ερώτημα, αίτημα του SND να προσθεθεί και το εξή ε, για την απόφαση για τον Jugendamt. Αρχικά να του καλέσουμε εκπρόσωπο τη Jugendamt στη μελλοντική συνεδρίαση τη Επιτροπή για να ακούσουμε και τη δική του οπτική και να στείλουμε και επιστολή ε, στον Επίτροπο. Εάν δεν υπάρχουν άλλες, ε, αν δεν υπάρχει κάποια διαφωνία, μπορούμε να το εγκρίνουμε. Ωραία, ευχαριστώ. Έχω και ορισμένες ανακοινώσεις. Να δω αν είναι εδώ ο ενδιαφερόμενος. Ωραία. Θα ήθελα όλοι να κοιτάξετε τον Λίο Κόξ. Και θα ήθελα να με κοιτάξει και εμένα ο Λίο Κόξ. Γεια σου Λίο. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Και πολύ χαίρομαι που όλοι σε κοιτάζουν αυτή τη στιγμή. Γιατί θα ήθελα εξ ονόματο της Επιτροπής Αναφορών να σε ευχαριστήσω που εργάστηκε σε αυτή την Επιτροπή εδώ και τόσο καιρό. Και όταν ήρθα μου είπαν ότι αυτό που δεν ξέρεις για τις αναφορές δεν αξίζει κανείς να τα γνωρίζει. Και εγώ έχω μάθει πολλά από σένα και ο Ντάνιελ ήσουν εξαιρετικά σημαντικός για το ΕΛΚ αλλά και για την ίδια την Επιτροπή. Τώρα μου είπαν ότι συνταξιδετούνται και οι νέοι πλέον. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Δεν ξέρω αν θα είσαι εδώ στην επόμενη συνάντηση, αν θα φύγεις πιο πριν. Και δεν ξέρω αν θα σε ξαναδούμε. Εάν ναι... Πάντα βεβαίως αυτό είναι ευχάριστο. Εάν όχι, να σε ευχαριστήσω εξ ονόματος της Επιτροπής και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την επόμενη και πολύ ωραία αυτή η περίοδο της ζωής σου. Ελπίζω να σου φέρει χαλάρωση, ξεκούραση, ε, ταξίδια, πολιτισμό, βιβλία, αθλητισμό, ό,τι θες. Ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις όμως, ελπίζω να το απολαύσεις. Ευχαριστούμε. and I also will come back to see. Και ελπίζω να έρθεις να μας ξαναδείς. Όταν πλέον δεν θα είσαι υποχρεωμένος να έρθεις, να έρχεσαι έτσι, εθελοντικά. Έχω και κάποιες ακόμα ανακοινώσεις συνδέονται με το περιβάλλον για να μειώσουμε τον όγκο χάρτου και με τους γενικότερους περιβαλλοντικούς στόχους ε, το τμήμα Β της μέσης διάταξης δεν θα εκτυπώνεται πλέον και θα είναι διαθέσιμο μόνο στο διαδίκτυο. Επιπλέον, και αυτό μπορεί να αφορά αρκετούς από εσά, ο αριθμός των αντιγράφων που θα περιέχουν το πρώτο τμήμα της μέσης διάταξης δηλαδή όλα τα ζητήματα που θα εξετάζονται στην Επιτροπή, έχει περιοριστεί σημαντικά. Τα μέλη μπορούν να έχουν ε, ένα αντίτυπο και ένας βοηθός μπορεί να έχει αντίτυπο. Αλλά στο προσεχές μέλλον θα δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τον, ε, την εκτύπωση φακέλων για τις συνεδριάσεις και κάποιες επιτροπές το έχουν ήδη κάνει με το λεγόμενο Paperless Committee. Όλα τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα ε, δείτε μέσω της εφαρμογής e-meeting. Και μετά το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση Frontex θα εκπονηθεί από κοινού από εμάς και από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ βάσει του κανόνα, δυνάμει του κανόνα 55. Αρχικά ε, η παρουσίαση του προσχεδίου θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου και η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 24 Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει το Φεβρουάριο και στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Στο επόμενο σημείο, από αριθμό 7, στα διάφορα, ο κύριος Μαριάς έχει ζητήσει κάτι για μια διαδικτυακή υπηρεσία ή πύλη. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ενημέρωσα πριν λίγο και τη συνάντησή μας των συντονιστών, ήθελα να ενημερώσω και την Επιτροπή μας ότι όπως όλοι γνωρίζετε η βασική προσπάθεια που κάνουμε είναι να είμαστε σε επαφή με τους ίδιους τους πολίτες, να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως την πρόσβασή τους στην Επιτροπή Αναφορών. Ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι με τα χρήματα που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχω διαμορφώσει μια πλατφόρμα διαβούλευσης και ενημέρωσης. Είναι το consultation.notismarias.gr. Είναι αυτή τη στιγμή μόνο στα ελληνικά αλλά θα είναι και σε άλλες δύο-τρεις γλώσσες εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί κανείς μέσα από αυτή την πλατφόρμα να συνδέεται απευθείας με την Επιτροπή Αναφορών. Έχει ένα ειδικό section «Ασκώ τα δικαιώματά μου», «I exercise my rights» και μπορεί κανείς μέσα από αυτή την πλατφόρμα να συνδεθεί με την Επιτροπή Αναφορών και την ηλεκτρονική φόρμα που έχει για να υποβάλει μια αναφορά στην Επιτροπή μας ή επίσης να υποβάλει μια καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Επίσης μέσα από αυτή την πλατφόρμα υπάρχει ένα link και συνδέεται με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί κανείς να δει μέσα από αυτό το link τη συνεδρίασή μας ζωντανά. Όπως ξέρετε η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσα από το link του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε έτσι μέσα από αυτή την πλατφόρμα μπορεί κανείς να δει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και αυτό να παραμείνει εκεί για να έχει κανείς μια εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ ως Ευρωβουλευτής να ενημερώνω τους πολίτες στην Ελλάδα για τους να μπορούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις μας οι οποίες βέβαια δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν σημαντικά θέματα και φαντάζομαι το μεσημέρι τρίτο που θα συνεδριάσουμε στις 3 η ώρα για τα θέματα των ε, υποθηκών στην Ισπανία, τα δικαιώματα των πολιτών, τις εξώσεις που υπάρχουν εκεί, θα είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και για τους Έλληνες πολίτες, γιατί τους απασχολούν και αυτά τα θέματα. Επομένως, θα σας στείλω και το link αυτής της πλατφόρμας και απλά ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή μας ότι υπάρχουν τρόποι μέσα από αυτά τα ποσά που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια άμεση επαφή με τους πολίτες και να περάσουμε σε μια μορφή ηλεκτρονικής δημοκρατίας, γιατί μέσα από αυτή την πλατφόρμα μπορεί κανείς να συμμετέχει σε φόρουμ, σε συζητήσεις, σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας κάποια στιγμή να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now I'm Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσουμε τον Χωσέ Ρικέλμεν Λόπεθ ε, εκ μέρους της Ένωση ε, των Θυμάτων τη Θαλιδομήνη στην Ισπανία. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ, αν μπορείτε να τηρήσετε και το χρονικό όριο. <clears throat> Hola, buenos días. Καλημέρα σα. Λέγομαι Χωσέ Ρικέλμε, είμαι πρόεδρο των ε, θυμάτων των Θαλιδομήνη και είμαι τον κύριο Βαστερετσέα που είναι αντιπρόεδρο. Για τι ερωτήσει που θα κάνετε. καταρχά θέλω να σα ευχαριστήσω όλου για τη συμμετοχή σα και στήριξη αυτήν την Επιτροπή Χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε αυτή τη συνάντηση και μάλιστα τόσο σύντομα. Σας ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι από πρώτο χέρι αυτό που θα σας παρουσιάσω σήμερα, 60 χρόνια μετά τα γεγονότα, αυτό που είναι γνωστό ως η τραγωδία της Θαλιδομίδης. Αυτή η χημική ένωση δημιουργήθηκε το 1954 χάρη στη γερμανική φαρμακευτική Grünenthal. Ήταν χάπια να κοιμηθεί κανείς να ηρεμήσει και ε, αντικαθιστούσε τα βαρβιτουρικά που πολλοί τα φοβούνταν. Ήταν πολύ σημαντική ανακάλυψη. Θέλαν τόσο να βγει στην αγορά που ξέχασαν να κάνουν τους ελάχιστους ελέγχους ασφάλειας και τις κλινικές δοκιμές. Και άρχισε να απολύται ως ένα καταπληκτικό ε, κατευναστικό και καταπολεμούσε και τις ναυτίες και τους εμετούς των εγγύων. Και μετά από 7 χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται τα αποτελέσματα μιας ε, ελλειπούς ή αν όχι παράτυπης ε, διαδικασίας ελέγχου από, το, ε, από την επιχείρηση αυτή και τις γερμανικές αρχές. Άρχισαν να εμφανίζονται παιδιά χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, με τρομερές τρευλώσεις και επίσης άλλες τρομερές αδυναμίες και αναπηρίες στα, στην, στην όραση, την ακοή, ε, τη γενετική και ε, ουροπητική λειτουργία, το, του, τα νεφρά και το πεπτικό σύστημα. Τα θύματα της θαλιδομίδης είναι γύρω στις 50.000 και στην Ισπανία ήταν 5.000 και γεννήθηκαν μεταξύ 61 και αρχών 62 και αποσύρθηκε σε όλες τις χώρες εκτός από την Ισπανία. Σε όλες ε, τις χώρες είχαμε αυτά τα τρομερά αποτελέσματα εκτός από τις ΟΠΑ που ποτέ δεν επέτρεψε να πολιθούν γιατί θεωρούσε ότι δεν είχαν υποστεί τα φάρμακα αυτά, τους αναγκαίους έλεγχους. Και χάρη στη δράση της υπαλλήλου Francis Kelsey, της ε, υπηρεσίας φαρμάκων των ΗΠΑ που θεωρείται ηρωίδα στη χώρα της, σώθηκαν χιλιάδες ε, βρέφοι στις ΗΠΑ. Τα περισσότερα κράτη, εκτός από την Ισπανία, δέχτηκαν την ευθύνη τους και έδωσαν βοήθειες οικονομικές και επιδόματα για να επιβιώσουν και να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα αυτά τα όντα σε συνθήκες αξιοπρέπειας και με καλυπτόμενες ανάγκες τους. Όλοι καθόρισαν μέσω νόμων ελάχιστες συντάξεις και οικονομικές βοήθειες στα θύματα ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας που άρχισαν να πληρώνονται στα τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετία του 70. Αυτές οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα αυξάνονται ανάλογα με τον πληθωρισμό και σε πολλές περιπτώσεις Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. βελτιώνονται σταδιακά μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, δυστυχώς, ε, είμαστε εδώ γιατί στην Ισπανία δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι έγινε στην Ισπανία όπως και στις άλλες χώρες. Και στην Ισπανία το Grünenthal πουλούσε αυτά τα φάρμακα και εξακολουθεί να έχει έδρα αυτή η εταιρεία και ε, ε, εργαστήρια στη χώρα μας και είναι πολυεθνική φαρμακευτική που έχει παγκόσμια δραστηριότητα. Όμως ε, στην Ισπανία εξακολούθησε ε, να πουλιέται ε, η θαλιδομίδη μέχρι το 1978. 16 χρόνια λοιπόν μετά την απόσυρσή της από την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρά το ότι ήταν γνωστά τα τρομερά, ήταν γνωστές οι τρομερές παρενέργειες, δεν υπήρξε νομοθεσία που να την απαγορεύει μέχρι το 1985. Τα θύματα στην Ισπανία ε, που υπολογίζουμε ότι ήταν 3.000 από τους οποίους ε, ζουν ακόμη μόνο 1.000 ε, υπολογίζουμε δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση και κανένα επίδομα. Τα περισσότερα θύματα χρειάστηκε να βασιστούν στις οικογένειές τους, στην εκκλησία, στη φιλανθρωπία ή ακόμη και στη ζητιανιά πεσμένη στους δρόμους των Ισπανικών πόλεων. Το 2015, 60 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε γιατί και δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Η ιστορία μας είναι παράλληλη με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εντελώς αντίθετη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει προς τα μπροστά με ρυθμό για να γίνει μια σύγχρονη ε, κατάσταση συνοχής, ενώ τα θύματα της ε, θαλιδομίδης είναι ακόμη ξεχασμένα, αποκλεισμένα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη μοίρα τους. Ήρθαμε εδώ να ζητήσουμε τη βοήθησά σας, να σας παρακαλέσουμε να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτή η τρομερή διάκριση που ε, υφιστάμεθα λόγω του ότι γεννηθήκαμε έτσι. Διακρίσεις ε, που είναι σε βάρος μας και που είναι πολύ διαφορετική η κατάστασή μας από όλα τα άλλα θύματα της θαλιδομίδης. Θέλουμε να υπάρξει κατανόηση. Γιατί δεν μας βοηθάει το Ισπανικό κράτος να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ακόμη και κυρώσεις, ούτω ώστε να επιτύχουμε το κράτος μας, το Ισπανικό κράτος, να αναλάβει την ευθύνη τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι η Θαλιδομίδη χρησιμοποιήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο για να αλλάξουν οι νόμοι και οι κανονισμοί για τον έλεγχο των φαρμάκων. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία για την παρακολούθηση και ασφάλεια αυτών των προϊόντων. Και χαιρόμεθα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα οργανώσει μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια αυτών των νόμων. Θέλουμε κάθε φάρμακο που λαμβάνει οποιοδήποτε να είναι ασφαλέ. Και αυτό χάρη στην καταστροφή τη Θελτομίδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωριστεί η περίπτωσή μα. Γιατί παρόλα αυτά μα έχει ξεχάσει η Ισπανία για τόσα χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε την κρίση με τα αγκούρια το 2011 που κόστησε στην Ισπανία 200 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα. Η υποψία, μόνο η υποψία της ε, Γερμανίας σήμαινε για τη χώρα μας απώλειες ένα δις. Πόσο έχει κοστίσει, πόσο θα είχε κοστίσει η κάλυψη των αναγκών της Θαντιδομίδης, τι θα είχε συμβεί στην Ευρώπη αν ένα ισπανικό εργαστήριο είχε κάνει κάτι αντίστοιχο για Γερμανούς Θέλουμε ένα μέλλον με αξιοπρέπεια για να καλύπτονται οι βασικές μας ανάγκες. Μέχρι ε, τη λήξη της υπόλοιπης ζωής μας. Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε. Χαιρόμεθα που μας υποστηρίζετε ομόφωνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να βοηθήσετε συγκεκριμένα τα θύματα στην Ισπανία για να ε, αναγνωριστεί ότι είναι άδικη η στάση της χώρας μας. Στόχος μας δεν είναι να υπάρξουν ε, ε, υπεύθυνοι. Θέλουμε να υπάρξει κοινωνικό διάλογο και ευαισθητοποίηση. Τέλο, επαναλαμβάνω ότι σα ευχαριστούμε όλοι που μα βοηθάτε στην πρόσβασή μα προ τα θεσμικά όργανα. Πρέπει επιτέλους ε, να υπάρξει αίσιο τέλο στην προσπάθειά μα. Είμαι πεπισμένος ότι με την βοήθειά σα θα υπάρξει σύντομα λύση. Γιατί σιγά σιγά τα θύματα στην Ισπανία πεθαίνουν. Γιατί έχουν περάσει 60 χρόνια και σε αυτά τα 60 χρόνια δεν έχουν δει ακτίνα ελπίδας. Η πολιτική είναι καλό, είναι πολύ θετικό να ε, βοηθήσετε σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι θα γραφτεί μια καλή σελίδα της ιστορίας Ευρώπης ε, προς την υποστήριξη των συμφερόντων και της ισότητας των πολιτών όλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να στραφώ τώρα στην Επιτροπή. Φλόριαν Σμιτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Α, τώρα σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η Θελιδομίδη σίγουρα είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές ε, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα στην Ευρώπη. Όπως πολύ σωστά είπε και ο αναφέρον, συνδέεται με τραγικό τρόπο και με την ύπαρξη και θέσπιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας γιατί ήταν ένας από τους κινητήρους μοχλούς σε ό,τι αφορά την ε, εναρμόνιση της ε, αδειοδότησης ε, των φαρμάκων πριν από 50 χρόνια. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως και κατανοούμε τις αξιώσεις του αναφέροντος και την κατάσταση στην Ισπανία που είναι ιδιαίτερη σε σύγκριση με άλλα κρατημέλη. Ωστόσο, υπάρχει και ένα μια νομική πτυχή ως προς την αναφορά και ένα πολιτικό σκέλος. Για το νομικό σκέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει στο παρελθόν σε μια σειρά ερωτήσεων και από τους ε, ευρωβουλευτές και πάντα υπενθυμίζαμε ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων των Ταμείων Αποζημίωσης και Υποστήριξης των Θυμάτων είναι ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ περιορισμένη επιρροή. Σε, αυτό, σε ό,τι αφορά λοιπόν το νομικό σκέλος, από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει κανείς εξ ονόματος του αναφέροντος. Για το πολιτικό σκέλος τώρα, γνωρίζουμε ότι πολλοί ευρωβουλευτές έχουν συναντηθεί στο παρελθόν με θύματα της Θαλιδομίδης και τους ε, στηρίζουν ενεργά και απέναντι στην εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας και μπορώ να πω ότι ο κύριος Ανδρεοκάητης πρόσφατα ο Αρμόδιος Επίτροπος δηλαδή, πρόσφατα συναντήθηκε με εκπροσώπους ε, των θυμάτων ε, της Θαλιδομίδης από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τον Ηνωμένο Βασίλειο για μια ανταλλαγή απόψεων και όπως είχε γίνει και προηγουμένω από τον Επίτροπο Μπόργκ, τον προκατοχό του. Υπάρχει λοιπόν και ένα πολιτικό σκέλος, όμως οικονομικής άποψη, καθαρά και μόνο, πολύ λίγα μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now I open the floor. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη. Κύριε Μαχτά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, αναφέροντα για την παρουσίασή του. Είδαμε και τις εικόνες. Κατανοώ το αίτημα που κάνατε, δηλαδή ότι δεν θέλετε να ενοχοποιήσετε κάποιον, βεβαίως, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει. Εσείς θα πρέπει να βρείτε τον ε, κατάλληλο τρόπο που θα γίνει αυτό. Εγώ δεν είμαι δεν έχω λάβει τέτοια νομιμοποίηση για να σας πω με ποιον τρόπο θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση, γιατί είναι απαράδεκτο τα θύματα να πληρώσουν δύο φορές. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις αναπηρίες που έχουν υποστεί και δεύτερον, από τον αντίκτυπο στην κοινωνική του ζωή. Και πολύ ωραία μας δείξατε και την πραγματικότητα της καθημερινής ζωή των ε, θυμάτων στην Ισπανία, χωρίς να στιγματίζουμε κανέναν. Κοιτάξτε, λέει και η Επιτροπή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει, αλλά τι κάνει εδώ πέρα αυτή η αναφορά τότε. Μπορούμε κάτι να προτείνουμε, να ασκήσουμε πιέσει, ούτω ώστε και εμεί ω ευρωβουλευτέ ε, ε, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση στην Ισπανία ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ω έχει. Και εγώ θα πρότεινα, βεβαίω προ συζήτηση το θέτω, να ζητήσουμε από το Ισπανικό κράτο να διοργανώσει μία συζήτηση με του ενδιαφερομένου, ενδεχομένω και με το ε, εργαστήριο Γκρούνενταλ, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση. Διαπραγματεύσεις λοιπόν μεταξύ της Ισπανίας, του Ισπανικού κράτους, ε, του Συλλόγου των Θυμάτων και του εργαστηρίου Γκρούνενταλ για να βρεθεί μία λύση, μία συμφωνία που να τους ικανοποιεί όλους, ούτως ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές τα θύματα αυτή την κατάσταση. Πρέπει και εμείς λοιπόν κάπως να πιέσουμε για να υπάρξει μια τέτοια διαπραγμάτευση με μια συμφωνία ωφέλιμη για όλους. Ευχαριστώ, Μάγκρετ. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την παρουσία σας εδώ. Ομολογώ ότι το σκάνδαλο αυτό είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι μας περιγράψατε εσείς. Ξέρω ότι και στην Ισπανία έχουμε πολλά θύματα, αλλά και στη Σουηδία. Με τον άνθρακα στη Σουηδία τη δεκαετία του 60 είχαμε πάρα πολλά θύματα και στη Γερμανία ξέρετε τι έχει γίνει και τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι ε, ε, ε φαρμακοβιομηχανίες προσπαθούσαν να πιέσουν, ε, να εκβιάσουν και να υπονομεύσουν. Και μόνο στη ΣΥΠΑ κατάφεραν κάτι να κάνουν ως προς αυτό. Αλλά Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι το τελευταίο σκάνδαλο. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και συνεχίζεται. Εδώ έχω αυτό το βιβλίο «Θανάσιμα φάρμακα και οργανωμένο έγκλημα» και στην Ισπανία κυκλοφορεί, υπάρχει στην αγορά εδώ και ορισμένα χρόνια. Υπάρχουν όλα τα ονόματα εκεί πέρα, όλα τα στοιχεία. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα τη Θελιδομίδης για να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μα παρουσιάσει τι ακριβώ έχει γίνει σε αυτέ τι χώρε. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ. Πάει αυτό, πέρασε. Είναι πολύ ωφέλιμο. Μα λένε μάλλον ότι πέρασε, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τα θέματα είναι ακόμα εκεί. Και για άλλα φάρμακα έχουμε δραματικέ επιπτώσει και παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη υγεία και το καθεξής και η μεγάλη φαρμακοβιομηχανία είναι από, τις πλέον δραστήρι, από τους πλέον δραστήριους κλάδους βιομηχανίας στην TTIP αυτή τη στιγμή και πρέπει και εμείς ε, να φροντίσουμε να μην υπονομεύεται η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί εδώ παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, θα μπορούσατε να μας κάνετε μια σύνοψη, μια παρουσίαση πότε σταμάτησε η παροχή αυτού του φαρμάκου, πότε και τι αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί στα θύματα τους ασθενείς. Γιατί νομίζω ότι η περίπτωση τη Ισπανίας είναι ένα παράδειγμα, αλλά δεν είναι μοναδική περίπτωση. Και εγώ πραγματικά αγανακτώ όταν βλέπω πώς η Grunenthal ενήργησε και οι εταιρείε που συσχετίζονται με την Grunenthal, τι έχουν κάνει. Πρέπει να μπουν στη φυλακή όλοι αυτοί για τα όσα έχουν κάνει. Και τα γνώριζαν, τα γνώριζαν. Και απλώς συνέχιζαν δωροδοκούσαν τους γιατρούς. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Πότε σταμάτησε η κυκλοφορία αυτού του φαρμάκου, ποιε αποζημιώσει υπήρξαν, σε ποιε χώρε. Γιατί η Γκρούνταλ ποτέ δεν πλήρωσε για ό,τι έκανε. Ευχαριστώ. Ελεονόρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, αναφέροντα που μας έφερε σήμερα εδώ το θέμα αυτό. Εγώ εδώ και μήνες από όταν ε, δηλαδή γνώρισα την ε, Ιταλική Ένωση Θυμάτων της Ταλιδομίδης έχω ασχοληθεί με το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι οργανώθηκε και συνέντευξη τύπου τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, στο Κοινοβούλιο όπου ε, εκφράστηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων απολύτως υπέρ μιας λύσης ε, του προβλήματος που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα τα οποία είναι θύματα φαρμακευτικού ε, σκανδάλου απερίγραπτου εύρους. Όπως είπε και η Μαργρέτε προηγουμένως, τα συμφέροντα των φαρμακευτικών ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλα, ήταν τεράστια ε, και επομένως έκρυψαν ένα σωρό πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος βέβαια να πούμε ότι και η γερμανική κυβέρνηση ε, έκρυψε κάτω από το χαλί πολλά πράγματα γιατί στη διάρκεια της διαδικασίας προσπάθησε με ταχύτητα να κλείσει την διαδικασία ούτως ώστε να αποφύγει ε, αναγνώριση αποζημιώσεων όχι μονάχα στα ε, θύματα του φαρμάκου στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες ε, της, Ευρωπαϊ... της Ευρώπης. Άρα είναι πολλά τα άτομα τα οποία δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση. Εδώ ας πούμε σκέφτομαι τα θύματα της θαλιδομίδης στην Ιταλία που ε, καμία αναγνώριση της κατάστασής τους ε, δεν έχουν επιτύχει, που δεν αφορούν μονάχα την καταστροφή που έχει προέλθει από την χρήση αυτή του, του σκευάσματος αλλά και ε, της μεγάλης καταστροφής της προσωπικής τους ζωής, ε, της υγείας τους ε, που αφορά όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Χρειάζονται βοήθεια και δεν την έχουν. Με την Ιταλική Ένωση Θυμάτων Θαλιδομίδης προσπαθούμε ε, να κάνουμε ε, κάτι παραπάνω, ε, να καταλάβουμε δηλαδή την πραγματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες των θυμάτων που ζουν με αυτά τα προβλήματα σήμερα. Ε, γιατί δεν αναγνωρίστηκε το πρόβλημά τους, δεν αναγνωρίζονται ως ανάπηροι ε, και δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση, άρα δεν έχουν και δυνατότητα ε, να λαμβάνουν οποιαδήποτε στήριξη και βοήθεια στην καθημερινή τους ζωή, στην καθημερινότητά τους. Επίσης, Θυμίζω ότι έχει ε, σταλεί και επιστολή από πολλές πολιτικές ομάδες ε, και από τη δική μου, το, θα τέλει του προηγούμενου έτους, μέσω της οποίας ζητούμε από την καγκελάριο Μέρκελ να ξανανοίξει τη συζήτηση ε, και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να βοηθηθούν τα θύματα την 7η Ιουλίου γνωρίζω ότι ε, υπήρξε μια συνάντηση θυμάτων της Θαλιδομίδης με την γερμανική κυβέρνηση και επομένως ελπίζω ότι κάπου θα καταλήξει αυτή η διαδικασία και επομένως θα έχει καλές επιπτώσεις και για τα θύματα της Θαλιδομίδης στην Ισπανία. Ε, βεβαίως εμείς ε, δεν έχουμε τέτοιου είδους αρμοδιότητα, πρόκειται για αρμοδιότητα αποκλειστική ε, των κρατών μελών. Ε, απ' την άλλη πλευρά όμως, μέσω ήπιας πίεση, soft power, θα μπορούσαμε να πιέσουμε κι εμείς έτσι ώστε αυτό το ζήτημα, το τόσο σημαντικό, να αντιμετωπιστεί με δύναμη, με διαφάνεια και οπωσδήποτε μέσα σε ένα πνεύμα δικαίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για την παρουσία τους εδώ και για την ενημέρωση που μας έκαναν. Είμαι συγκλονισμένος με αυτά τα οποία είδα και το δράμα όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Και θα πρέπει η Επιτροπή μας εδώ να ασκήσει κάποια πίεση, να υπάρξει μια απάντηση στο αίτημα των αναφερόντων. Διότι ο στόχος αυτής της Επιτροπής είναι να μπορεί να συνδράμει, να μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε οι αναφορές οι οποίες έρχονται να έχουν και κάποιο πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι προφανές ότι πρόκειται για μια τεράστια ευθύνη της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας και δεύτερον ότι δεν έχει γίνει υπάρξη αποζημίωση μέχρι στιγμής και ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα έχει διάσταση ευρωπαϊκή, έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή μας, παρότι φαίνεται ότι από πρώτης πλευράς ματιάς δεν έχει διότι όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την χάρτα των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει στη συνθήκη της Λισαβόνας μία από τις βασικές αρχές είναι να υπάρχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα και αποτελεσματική δικαστική προστασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προφανές ότι τα θύματα αυτά είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι στιγμής δεν έχουν την αποτελεσματική δικαστική προστασία. Το ερώτημα είναι πού θα έχουν αυτή τη δικαστική προστασία και με ποιο τρόπο. Αν θα την έχουν στα ισπανικά δικαστήρια όπου εκεί θα πρέπει να ασκήσουν την αγωγή αποζημιώσεως ενάντια σε αυτούς που φταίνε βεβαίως, σε αυτούς που έχουν την ευθύνη, δηλαδή στην συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία ή εάν θα πρέπει να στραφούν οι ίδιοι στα γερμανικά δικαστήρια, ούτως ώστε να έχουν αυτή την προστασία. Επομένως το πρώτο ζήτημα που πιστεύω θα μπορούσε να μας βοηθήσει η Επιτροπή είναι να έχουμε μια καταγραφή της υπόθεσης. Πόσες χιλιάδες θύματα υπάρχουν, αν έχουν δοθεί αποζημιώσεις μέχρι στιγμής, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και πού είναι η αρμοδιότητα, σε ποιο χώρο, σε, ποιο, σε ποια σε ποιο κράτος πρέπει να ασκηθεί αυτή η αγωγή αποζημιώσεως και πού βρισκόμαστε. Άρα εδώ θα μπορούσε να συμβάλλει η Επιτροπή, εννοώ η Κομισιόν, και η δική μας Επιτροπή να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Πρώτον, ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ούτω ώστε το άμεσο δικαίωμα των πολιτών, των θυμάτων για προστασία δικαστική να έχει ένα αποτέλεσμα που αυτό συνεπάγεται προφανώς και μια αποζημίωση. Και δεύτερον, συμφωνώ με τον συνάδελφο από τη Γαλλία που έθεσε το ζήτημα της πίεσης για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα ζητήματα. Επίσης, όπως είπε και η συνάδελφος Ήβη, υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο, αυτό του soft power, δηλαδή της πίεσης σε ένα επίπεδο προς την γερμανική κυβέρνηση για να υπάρξει μια προστασία, να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, μια αποζημίωση σε αυτά τα χιλιάδες θύματα που από ό,τι καταλάβα δεν είναι μόνο στην Ισπανία, είναι και σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες να βοηθήσει η Επιτροπή μας, πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά, πρέπει να έχουμε αυτές τις ε, εκθέσεις από πλευράς της Κομισιόν και να δούμε παραπέρα πώς μπορούμε εμείς πρακτικά να συνδράμουμε στη στήριξη των αναφερόντων και να μην μείνει απλά μια συζήτηση καλών προθέσεων και συμπάθειας στους ίδιους τους αναφέροντες. Πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Now, Rosa, the floor το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον ε, Χωσεν Λόπεθ, Ρίκελ Μελόπεθ και το Ραφαέλ εκπροσωπούν πολλούς και νομίζω ότι μας έκανε ένα μάθημα αγώνα και αξιοπρέπειας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αναφορών ως ε, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας στηρίζουμε για να επιτύχετε τον τελικό σας στόχο, τη δικαιοσύνη. Να μην υπάρχουν διακρίσεις και μεταξύ των θυμάτων και όλα τα θύματα της Θελδομίδης να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ξέρουμε ότι είναι ιστορική σημασία η ιατρική τραγωδία. Δεν είναι μόνο ισπανικό, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, πολιτικό και ανθρωπιστικό. Αυτό θα πρέπει να ενώσει όλες τις κυβερνήσεις, όλους τους εκλεγμένους για να υπάρξει δίκαια λύση. Είναι απαράδεκτη, εξευτελιστική αυτή η κατάσταση στην ε, Ισπανία δεν έχουν αναγνωριστεί παρά μόνο πολύ λίγα θύματα της ε, θαλιδομίδης και σιγά σιγά βέβαια αποβιώνουν γιατί έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια. Άρα είναι επίγον να βρεθεί λύση για να βοηθήσει, να βοηθήσει, να ανακουφίσει τόσο πόνο. Και εσείς είπατε ότι είναι σαν ολοκαύτωμα η τραγωδία της θαλιδομίδης και συμφωνώ. Οπότε βασίζομαι στην πρόταση που έγινε από τον πρώτο ομιλητή, η Επιτροπή μας δηλαδή, να ζητήσει να γίνει κάποια να αναλυφθεί κάποια πρωτοβουλία για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι στις 23 ε, Σεπτεμβρίου θα το συζητήσει το θέμα αυτό το ε, αστικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, να δούμε πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση η ομάδα μας θα κάνει ό,τι μπορεί και μέσω της Επιτροπής Αναφορών, ούτω ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα, να το ξεμπλοκάρουμε, γιατί ε, πρέπει να αντιμετωπιστείτε όπως τα υπόλοιπα θύματα σε όλες τις άλλες χώρες, χώρες της Ευρώπης. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να είναι θύμα της ταλιδομήτης, Εγώ ενήθηκα το 1965 τότε που γιόταν ακόμη αυτό το φάρμακο. <clears throat> Άρα πρέπει να πω ότι απαιτείται δικαιοσύνη, είμαστε στο πλευρό σας, έχετε όλη τη στήριξη της ομάδας μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. <clears throat> Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε τη στήριξη όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρη, συγγνώμη. Θα έχετε τη στήριξη όλων μας. Δύο λόγια να πω μονάχα. Είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις στην Επιτροπή Αναφορών και όλες οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν να σας ακούσουν και να μοιραστούν απόψεις μαζί σας. Ε, ε, πραγματικά είναι μια προσπάθεια η οποία έχει γίνει από όλες τις πολιτικές ομάδες και από το σύνολο της ε, Επιτροπής Αναφορών που σας στηρίζει. Ο Κάρλ, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ερμηνεύσω κατά κάποιο τρόπο τη σκέψη του ΕΛΚ. Εδώ η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι δύσκολη. Ξέρετε, εγώ είμαι βιοχημικός και μετά από το τέλος των σπουδών μου στην βιοχημία έκανα έρευνα για ε, χημικά ε, χημικά συστατικά και ουσίες και πραγματικά ε, σας λέω λόγω αυτής της ε, εμπειρίας μου ότι η θαλιδομίδη δεν έπρεπε ποτέ μα ποτέ να χορηγηθεί σε ανθρώπους. Είναι πραγματικά έγκλημα και συμφωνώ, μαζί, συμφωνώ με όσους είπαν ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση και στην Κομισιόν και στην Ισπανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και να συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε. Ευχαριστώ Σολεδά. Ευχαριστώ. Και εγώ οπωσδήποτε βέβαια να καλωσορίσω και να εκφράσω όλοι μας την αλληλεγγύη <clears throat> όπως ε, είπατε και εσείς Πρόεδρε ο οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι θύμα αυτού του φαρμάκου. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της σύγχρονης ιατρικής. Ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα. Ήταν τεράστια τραγωδία, τεράστια καταστροφή. Έχουν αναφερθεί πολλά χαρακτηριστικά και έχει υποθεί ότι αυτό προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης. Ήτανε, χρειάστηκε δυστυχώς τέτοια τραγωδία για να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αναγκαία ανταπόκριση για όλα τα θύματα που δεν έχουν λάβει επαρκή βοήθεια, δεν έχουν λάβει δικαιοσύνη μετά από 50 χρόνια, δεν έχουν εισακουστεί τα αιτήματά τους. Πιστεύω δεν υπήρξε ποτέ η αναγκαία ελάχιστη πολιτική βούληση για να υπάρξουν οι αναγκαίες ε, νομικές λύσεις. Απλώς ε, έγιναν έρευνες για το τι έγινε. Ξέρουμε επίσης ότι καταστράφηκαν και διάφορα έγγραφα και υπήρξαν ε, συμφωνίες μεταξύ κάποιων χωρών και φαρμακευτικών εταιριών. Και τελικά εποφελήθηκε αυτή η εταιρεία με τέτοιο ξεδιάντροπο τρόπο από την κατάσταση αυτή που προκάλεσε. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αδικία. Βεβαίως δεν έχουμε νομική αρμοδιότητα για να σας χορηγήσουμε αποζημιώσεις, αλλά μπορούμε να εκφράσουμε την πολιτική μας βούληση. Ναι, μεν έχουν περάσει τόσε δεκαετίες, αλλά πρέπει να μελετήσουμε το θέμα αυτό, να κάνουμε την αναγκαία προσπάθεια έρευνας, να δούμε τι συνέβη όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά σε όλη την ε, Ένωση και είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι πρέπει να το κάνουμε αυτό για να στηρίξουμε τα αιτήματά σας τόσο στην Ισπανία αλλά και αυτά που εκκρεμούν ακόμη στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Βεβαίως στην Ισπανία το 2010 υπήρξε ένα διάταγμα που προσπαθούσε να υπάρξει αναγνώριση των θυμάτων. Ήταν η πρώτη τέτοια αναγνώριση στην Ισπανία και βεβαίως και η Ένωση Θυμάτων στην Ισπανία τη θεωρεί ανεπαρκή αυτήν την ρύθμιση. Να γράψουμε λοιπόν στην Ισπανική κυβέρνηση για να καθίσουν μαζί με αυτήν την ένωση να υπάρξει ένας διάλογος, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το διάταγμα που όπως είπα η Ένωση θεωρεί ότι είναι πολύ περιοριστικό και δεν έδωσε ούτε την αναγνώριση ούτε τις αναγκαίες αποζημιώσεις. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου πρόταση. Δεύτερον, υπόθηκε ότι δεν έχουμε καμία νομική αρμοδιότητα, αλλά εάν υπάρχει η πολιτική βούληση, όπως είπε και ο αρμόδιος επίτροπος για την υγεία στην τελευταία παρέμβαση που έκανε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είπε ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Και προσφέρθηκε να μελετήσει την υπόθεση. Σημαντικό πιστεύω να του αποστείλουμε ένα ερώτημα ως Επιτροπή στον Επίτροπο Υγείας, να δεχθούμε το αίτημά του, να ασχοληθεί, να μας πει τι μέτρα, τι απάντηση τι θα μπορούσε γενικά να κάνει για να υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό νομίζω χρειάζεται η Ένωση αυτή και οι πολίτες μας. Και τρίτον, αυτή η μελέτη στην οποία αναφερθήκαμε είναι και αυτή πολύ σημαντική. Να υπάρξει λοιπόν η αναγκαία έρευνα. Θα καλούσα και την νομική επιτροπή, παρά το δεν έχουμε νομική αρμοδιότητα, θα ήθελα να ακούσω και μια νομική άποψη της Επιτροπής Νομικών Εποθέσεων του Κοινοβουλίου για να δούμε σε τι βαθμό μπορεί να υπάρξει από το συγκεκριμένο κράτος μέλος και νομική αντίδραση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ μάλιστα που κάνατε και συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Κυρία Σαλίνα. Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά ε, καλώς ήρθατε Χωσέ και Ράφα. Δυστυχώς χρειάζεται να έρθετε πολλές φορές. Ε, ξέρετε πόσο με θλίβει το να ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά υπάρχει ένας χάρτης ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άμα δεν χρησιμεύει ούτε γι' αυτό, τότε είναι στα λόγια μόνο. Εκεί μιλάμε για το δικαίωμα στην υγεία, για το γεγονό ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις για λόγους ε, εθνικότητας και ότι υπάρχει δικαίωμα σε βοήθεια και σε κυρίως προστασία της υγείας όπως είπα. Συμφωνώ να υπάρξει έκθεση και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ναι μεν στην Ισπανία 16-12 υπήρξε αυτό το βασιλικό διάταγμα που έδινε αναγνώριση και έδινε κάποια επιδόματα, κάποιες κοινωνικές παροχές αλλά όχι πλήρη αποζημίωση και υπήρχε προθεσμία μόνο ενός μηνός για να υποβάλει κανείς αίτημα, να αναγνωριστεί ως αίτημα. Άκουσα τους ε, εκπροσώπους ε, του κυβερνητικού κόμματος εδώ που ε, να θυμίσω ότι υπήρξε και μια συνέντευξη τύπου στις 27 Μαΐου όπου ήταν και ο Υπουργό Πόνς Υγείας λέγοντας ότι θα κάνουν, θα κάνουν ό,τι μπορούν αλλά σας παρακαλώ, σας παρακαλώ εάν έχετε όντως πολιτική βούληση κύριοι του κυβερνητικού κόμματος ε, συνεργαστείτε με την Ένωση καθίστε επιτέλους στο τραπέζι σας περιμένουμε, σας περιμένουμε λίγη η θητεία σας η πρώτη δεν αρκούν τα λόγια έχουν περάσει τόσα χρόνια Δυστυχώς, λίγοι έχουν απομείνει ζωντανοί. Τι περιμένετε. Αναφερθήκατε στην κρίση για τα αγκούρια. Υπήρχε μια υποψία και γι' αυτό έχασε τόσα λεφτά η, η Ισπανία. Ξέρετε ε, πόσους πόρους έχει 11 δις δαπανά για τέτοιους σκοπούς η Καθολική Εκκλησία. Δεν μπορούμε να βρούμε πόρους να βοηθήσουμε τα θύματα ενός φαρμάκου χρειάστηκε να φτάσουμε ως εδώ. Ε, ήρθε η ώρα επιτέλους να πάρουμε μια απόφαση, να υπάρξει μια λύση. Γιατί τα θύματα αυτά όλη τους τη ζωή χωρίς να έχουν λάβει βοήθεια. Και νομίζω ότι όλα αυτά μας λένε κάτι πολύ κακό και για τη χώρα και για την Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Στέρι Κάμπρας. Και μετά θα πρέπει να κλείσει η συζήτηση. Α, και ο Πέτερ. Α, μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Φυσικά, Πέτερ, και εσύ. Μετά τον Πέτερ, θα κλείσω τον κατάλογο μιλητών γιατί πρέπει να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Τέρι Κάβρας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω συζητήσει μαζί σας, που είχα την τιμή να έρθω σε επαφή με ενό συστημάτων της Θαλδομίδης, όχι μόνο από την Ισπανία, και, αλλά και από άλλες χώρες. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου, απολύτως. Φυσικά είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, γιατί υπήρξαν θύματα στην ε, Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την ε, Σουηδία και βέβαια στη Γερμανία που φέρει ειδική ευθύνη. Αλλά οι αναφέροντες είναι Ισπανοί. Άρα θα ασχοληθώ, με την περίπτωση της Ισπανίας για να μην χανόμαστε και να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέμε και τι ζητάμε. Είναι σίγουρο, όπως είπε και η συνάδελφός μου, ότι η Ισπανική κυβέρνηση στις 6-8-2010 έβγαλε ένα διάταγμα. Αλλά κοιτάξτε, το έβγαλε Αύγουστο, ε. Να δούμε και τη χρονική στιγμή. Είναι απόλυτα, απόλυτα απαράδεκτο, είναι απίστευτο. Και επιπλέον, επιπλέον είναι κοινωνικά επιδόματα πρέπει να κάνουμε και τα εξή δύο. Πρώτα απ' όλα, αποζημιώσει. Είναι μερικέ εκατοντάδε θύματα. Έχουν απομείνει εκατοντάδε σε όλη την Ευρώπη στην πραγματικότητα, οπότε λιγότερο στην Ισπανία. Εύκολα μπορούν να αποζημιωθούν. Είναι σκανδαλώδε που δεν έχει συμβεί ακόμη. Δεύτερον, ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί, γιατί το Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα, αλλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κυρώσεις, δικαστικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα κατά εκείνων και εκείνων των διοικήσεων, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά της Ισπανικής διοίκησης, που συνέχισε να δίνει άδεια για την πώληση και χορήγηση του φαρμάκου, ενώ ήταν γνωστά τα τρομερά, ήταν γνωστές οι τρομερές παρενέργειες. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε αποζημιώσει και κυρώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πέτερ. Ευχαριστώ. Μια συμπλήρωση. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που είναι παρόντες και παρουσιάζουν το θέμα. Είμαι 59 ετών, ξέρετε. Στην Ανατολική Γερμανία δεν είχαμε πολλές περιπτώσεις. Γιατί ξέρετε υπήρχε αυτό το σιδηρούν παραπέτασμα και ούτως ή άλλως αυτά τα φάρμακα δεν ήταν διαθέσιμα. δεν ήταν απλώς τραγωδία πρέπει να πω, ήταν και έγκλημα. Τραγωδίες εντάξει, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αλλά αυτό εδώ συνέβη συνειδητά. Γιατί ήταν γνωστές οι παρενέργειες και συνεχίστηκε να δίδεται η άδεια, παρατάθηκε η άδεια. Και δεν έχουν τιμωρηθεί οι ένοχοι. Βεβαίως δόθηκαν αποζημιώσεις, αλλά πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Κοιτάξτε, είναι έγκλημα λοιπόν, τονίζω. Και βεβαίως ε, αντιμετώπισαν αδικίες και τα θύματα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έλαβα πληροφόρηση από τον βοηθό μου εδώ, τις 26 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα όπου ζητάει να υπάρχει ε, δίκαιη αποζημίωση για τα θύματα από τα σκάνδαλα φαρμάκων. Υπάρχει συγκεκριμένο ψήφισμα. Αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε. Από νομική άποψη μας λένε ότι η κατάσταση έχει ως έχει, αλλά πρέπει να επιμείνουμε από πολιτική άποψη. Βεβαίως για πολλά κράτη είναι δυσάρεστο αυτό, αλλά πρέπει να παραμείνει στην μέση διάταξη. Ξέρετε, παρά το ότι προσπαθούν να το καταχωνιάσουν. Πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε να μείνει στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να γράψουμε σε όλα τα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν θύματα, να τους πούμε ότι πρέπει να ασχοληθούν και νομίζουμε ότι το ψήφισμα αυτό μας δίνει την αναγκαία όθηση. Έχει ασχοληθεί ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας πούν τι συνέχεια έδωσαν στο θέμα αυτό, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ανεξάρτητα από τη σωματική βλάβη που δεν μπορεί να διορθωθεί, πρέπει να κάνει το ελάχιστο μια δημοκρατική κοινωνία για μια δίκαιη αποζημίωση. Αρμόζουσα. Εμείς ε, σας ευχαριστούμε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να δοθεί συνέχεια και στο ψήφισμα, όντως. Ε, τώρα θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο για δύο λεπτά στον εισηγητή, στον αναφέροντα, συγγνώμη, και παρακαλώ να μην ξεπεράσει τα δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους για την τιμή που μας κάνατε προσκαλώντας μας. Βεβαίως υπόθηκε ότι είναι πρόβλημα κρατών. Εδώ είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Θαλιδομίδη πήρε άδεια πώληση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Για τα θύματα στην Ισπανία ξέρουμε ποιες είναι οι τρεις άμεσες ευθύνες. Η πρώτη και η σοβαρότερη είναι της γερμανικής φαρμακευτικής Grünenthal που παρήγαγε απευθεία και μάλιστα πούλησε απευθεία στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Δεύτερον, οι γερμανικές αρχές είναι υπεύθυνε γιατί δεν έκαναν του αναγκαίου ελέγχου πριν εξαχθεί αυτό το φάρμακο και κατόπιν υπάρχουν άμεσες ευθύνε όλων των χωρών που επέτρεψαν την εισαγωγή και την ε, πώληση του φαρμάκου αυτού. Όπως είπε ο κύριος Τέρη Κάβρας, είναι ακόμη πιο σοβαρή η περίπτωση της Ισπανίας γιατί ήταν γνωστές οι παρενέργειες αλλά για λόγους έλλειψη ελέγχων ή γιατί υπήρχε τεράστια εμπιστοσύνη στο γερμανικό κράτος παρά το ότι λοιπόν υπήρχαν αυτές οι αμφιβολίες εξακολούθησε λόγω εμπιστοσύνης και φαίνεται ότι υπήρχε και στην Ιταλία τέτοια εμπιστοσύνη λόγω εμπιστοσύνης στο γερμανικό κράτος εξακολούθησε η χορήγηση αυτού του φαρμάκου. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θέμα πρώτης σημασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς ως ε, αναφέροντες. Ε, δεν ξέρουμε βέβαια τα διαδικαστικά, αλλά αν αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα τότε ποιο είναι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω με το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσοι ε, συμμετείχαν. Όπως ορθώς ε, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά κάποιο τρόπο εδώ υπάρχει το νομικό σκέλος και το πολιτικό σκέλος του προβλήματος. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι εδώ είναι ανθρωπιστικό κιόλας το ζήτημα. Μπορούμε να στείλουμε επιστολή στον ε, Υπουργό ε, Κοινωνικών Θεμάτων για να του ζητήσουμε να μας πει τι μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Επίσης, να κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση να αναλάβει δράση σε συνεργασία με την οργάνωση εκπρόσωπο της οποίας ακούσαμε σήμερα. Επίσης, ε, με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να μάθουμε τι μέτρα έχουν πάρει για το θέμα αυτό άλλες χώρες. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο ε, καλών πρακτικών και αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο. 16 ε, ε, χρόνια έχουν περάσει. 60 χρόνια έχουν περάσει από την απαγόρευση κυκλοφορίας ε, του φαρμάκου και σίγουρα πολλά έχουν γίνει, επομένως καλό είναι να ξέρουμε και υπάρχουν όπως γνωρίζουμε και ορισμένες χώρες μέλη που όντως έχουν δώσει αποζημιώσεις. Τρίτον, να στείλουμε επιστολή ε, στον ε, Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα υγείας. Τέταρτον, ε, να αναφέρουμε ε, στα, στις επιστολές αυτές ε, αυτό το ψήφισμα το οποίο ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο και το οποίο ορθώς ανέφερε ο Πίτερ προηγουμένως. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση, ε, αρκετή πίεση στις ισπανικές αρχές, στην ισπανική κυβέρνηση και οπωσδήποτε ε, θα το κάνουμε ε, και βεβαίως όπως άλλωστε είπαν και όλοι οι συνάδελφοι να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος γιατί να γράψουμε ε, στον ε, Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και όχι στον Υπουργό Υγείας. Α, είχα την εντύπωση, λέει η Πρόεδρος, ότι είναι ένα το Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα αποστείλουμε την επιστολή στην κυβέρνηση και δεόντως θα προωθηθεί. Ε, ναι, γιατί δεν είναι εδώ ζήτημα κοινωνικής, ας πούμε, αποζημίωσης ή κοινωνικού επιδόματος. Είναι θέμα αποκατάστασης δικαιοσύνης. Ναι, ναι, βεβαίω, έχετε δίκιο, λέει η Πρόεδρος, αλλά είχα την εντύπωση ότι είναι ένα το Υπουργείο. Από ό,τι μου λένε εδώ είναι το ίδιο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. <laughs> Κύριε Τερεκάμπρας, δεν ξέρετε τι γίνεται στη χώρα σας. Ναι, αλλά εγώ είμαι καταλανός όμως. <laughs> Εντάξει, τώρα αυτό το εξηγεί, είναι, είναι μια εξήγηση, αλλά όχι όμως δικαιολογία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε. Κύριε Μαρτάν, Αυτό που με προβληματίζει εδώ είναι η έλλειψη στόχευσης όσον αφορά την ευθύνη των εργαστηρίων Grünenthal. Γιατί έχω την εντύπωση ότι τη γλιτώνουν πάλι. Ε, πρέπει να πούμε ότι πρώτος υπεύθυνος είναι το εργαστήριο Grünenthal δεν έχω εδώ στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ζητήσουμε από την Κρινολίτα να μας πει τι είδους και τι ύψους αποζημιώσεις έχει δώσει μέχρι τώρα γιατί μπορεί να προκύψει ότι δεν έχουν πληρώσει δεκάρα τσακιστή. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια κατάσταση όπου ε, το εργαστήριο το οποίο ε, είναι υπεύθυνο δεν πλήρωσε τίποτα. Σε όλες τις άλλες ε, περιπτώσεις, περιβάλλον κλπ. λέμε ότι ο υπεύθυνος πληρώνει. Εδώ θα την βγάλει καθαρή χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρόεδρος, πολύ καλή ιδέα και ε, πραγματικά χαίρομαι γιατί με μεγάλη ρόμη αναφέρατε το, ε, την άποψή σας. Ε, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό που λέτε. Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Πολύ ωραία. Σας, ε, πρέπει να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές σας ευχαρίστησαν. Είναι η σειρά μου να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ, που μοιραστήκατε τον προβληματισμό σας μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Περνάμε στο επόμενο θέμα, ε, είναι η 717 του 2014 ε, για την κατάργηση της, ε, της διαφορετικής ώρας καλοκαιριθερινής μάλλον και χειμερινής ώρας 1934 και, και επίσης μια σειρά άλλων αναφορών με το ίδιο θέμα. Θα σας θυμίσω ότι ο Γιώργος Σουίν έχει γράψει ένα πολύ καλό, ένα πολύ ωραίο τραγούδι ε, για τη θερινή και την χειμερινή ώρα, on summer time, on winter time, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα δώσω αμέσως το λόγο στον Πίτερ Ντεμάγερ από την Επιτροπή. Good morning. This uh, chair. Uh, ε, καλημέρα κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν ε, την αίθουσα να το πράξουν ε, ηρέμος και ησύχω, ε, έτσι ώστε να προχωρήσουμε εμείς στις εργασίες της Επιτροπής μας. Κύριε Ντεμάιερ, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας δώσω ε, κάποια στοιχεία όσον αφορά τις οδηγίες. Ε, η οδηγία για την θερινή ώρα είναι αυτή η οποία ε, εισάγει την αλλαγή ώρας δίστου έτους. Τέλη Μαρτίου λοιπόν θερινή ώρα, τέλη Οκτωβρίου χειμερινή. Καλό είναι να γνωρίζει κανείς ε, ότι η Κομισιόν και ε, το Κοινοβούλιο δεν ε, πήραν απόφαση συλλογική για την αλλαγή της ώρας. Ε, ήταν αποφάσεις οι οποίες ήδη στη δεκαετία του 60 και 70 είχαν πάρει μεμονωμένες χώρες. Για πολλούς λόγους ε, τότε εισήγαγαν ε, την θερινή και χειμερινή ώρα τα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο τώρα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτό που συνέβη είναι ότι ανελήφθη το 81 πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν ε, που πρότεινε εναρμόνιση του ζητήματος ε, της ώρας στις διάφορες χώρες που την εφάρμοζαν ήδη έτσι ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά γιατί σας είπα τη δεκαετία του 60 και του 70 είχε ήδη εισαχθεί σε μερικές χώρες η θερινή ώρα και επομένως ε, κυρίως ε, ε, προέκυψαν προβλήματα, προέκυπταν μάλλον τότε προβλήματα στις διεθνείς μεταφορές και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρώτη πρόταση οδηγίες η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό έγινε για πέντε χρόνια αρχικά και μετά στην αρχή είχαμε ε, εναρμόνιση της αρχής και όχι του τέλους ε, του διαστήματος. Ε, μετά όμως είχαμε την ένατη οδηγία του 2000 μέσω της οποίας υπάρχει πλήρη εναρμόνιση το, της θερινής και της και της χειμερινής ώρας σε μόνιμη βάση πλέον και όχι πενταετία όπως πριν. Ε, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εναρμονισμένη προσέγγιση από όλες τις χώρες έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά και η εσωτερική αγορά. Δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα άλλο και ε, νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομος και ακριβής. Θα ήθελα να αναφέρω ότι οι επιτροπές ε, Γιούρι, Ίντρε και ε, Τραν ε, διοργάνωσαν κοινή εκδήλωση για αυτό το ζήτημα το Μάρτιο. Βλέπω ότι οι ορισμένοι συνάδελφοι δεν τους ξέρω μάλλον. Ο κύριος Σβόμποντα και μετά ο κύριος Ρόλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να με γνωρίζετε. Όχι. Ε, βεβαίως. Βεβαίως και σας γνωρίζω. Ναι, όπως είπατε, οι τρεις επιτροπές πράγματι έκαναν μια πολύ πετυχημένη ακρόαση στην οποία προσκαλέσαμε εκπροσώπους του κλάδου της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας. Εξετάσαμε ακόμα και νομικές πτυχές ε, της οδηγίας ε, του 2001, που ήταν η τελευταία. Το αποτέλεσμα της ακροάσης ή μάλλον να διακρίνουμε μεταξύ δύο στοιχείων. Πρώτον είναι η εναρμονισμένη προσέγγιση, είναι κάτι το θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι είναι κάτι σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε είναι κατά πόσο έχει νόημα σήμερα να αλλάζουμε από την ε, χειμερινή στη θερινή ώρα. Μήπως θα ήταν καλύτερο να έχουμε μία ώρα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ είχαμε παρουσιάσεις από τον κλάδο των μεταφορών, της ενέργειας και της υγείας. Η ενέργεια, οι μεταφορές και το καθεξής είπαν ότι εντάξει, ε, δεν υπάρχουν ούτε πλεονεκτήματα ούτε μειονεκτήματα της μίας ή της άλλης επιλογής. δεν υπάρχει λόγος για εκείνους για να αλλάξει η ώρα. Αλλά στον τομέα της υγείας, βάσει μελέτης από, σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, η γνωμοδότηση ήταν εξαιρετικά αρνητική. Ένας Γερμανός καθηγητής μας έδωσε στοιχεία για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ε, που δαπανώνται για αυτό το λόγο και αναφέρθηκε ότι το 80% των ε, πολιτών δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα την αλλαγή ώρας, ενώ το 20% αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Το 80% δεν μπορεί να κατανοήσει ότι αυτό το 20% αντιμετωπίζει πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν ε, σαφής διάκριση απόψεων για αυτό το θέμα. Ακούσαμε αντίδραση και της Επιτροπής στην ακρόαση. που ήταν ε, αρκετά έντονη, γιατί η Επιτροπή ουσιαστικά ανέφερε ότι έχει κάνει μελέτες που δείχνουν ότι κατά τη χρονική στιγμή υιοθέτησης της ε, οδηγίας υπήρχαν λόγοι να γίνουν αυτές οι αλλαγές της ώρας και ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να κάνει τίποτα ως προς αυτό το ζήτημα. Στη φάση της προετοιμασίας τώρα έχουμε προφορικό ερώτημα, το οποίο θα τεθεί μετά τις ε, καλοκαιρινές διακοπές. Προς την Επιτροπή θα τεθεί λοιπόν στην Ολομέλεια. ούτως ώστε η Επιτροπή να μας παρουσιάσει τα επιχειρήματά της για τη διατήρηση της αλλαγής της ώρας και μετά θα δούμε βάσει των απαντήσεων της Κομισιόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αν θα ζητήσουμε ψήφισμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Όμως, δεν αντιδρούμε παθητικά, κάτι γίνεται και υπάρχει σημαντικός αριθμός μελών του Κοινοβουλίου σε όλες τις πολιτικές ομάδες που στηρίζουν την κατάργηση των αλλαγών της ώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρούλ. Ευχαριστώ πολύ. Να αναφέρω μερικά επιχειρήματα ακόμη. Αυτό απασχολεί πολλούς χιλιάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνουμε επιστολές, αναφορές, ακόμη και στα κράτη-μέλη υποβάλλονται τέτοιε αναφορές και η Κομισιόν μας είπε πώς προέκυψε. Ενδιαφέρον πώς προέκυψε η θερινή ώρα δηλαδή. Αλλά κανείς δεν μας λέει συγκεκριμένα πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Ποια είναι η διαδικασία που θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν βέβαια αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποβάλουμε τους ανθρώπους δύο φορές το χρόνο σε αλλαγή ώρας. Οι λόγοι που υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν τώρα. Δεν έχουμε πλέον εκτίματα από πλευρά κατανάλωσης ενέργειας. Δεν έχουμε εξοικονόμηση. Και τα κράτη-μέλη λένε είναι αρμόδια η Ένωση και η Ένωση λέει το αντίστροφο. Υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον τότε η Επιτροπή υπέβαλε την οδηγία και τώρα αν θέλει μπορεί να υποβάλει μία αντίστροφη πρόταση. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν αυτή η πρόταση για να σταματήσει αυτή η παράλογη κατάσταση. Περιμένω μία απάντηση. Μήνες η Κομισιόν δεν μου δίνει σαφή απάντηση. Έγραψα στον Επίτροπο. Έχει λόγο λοιπόν. Έχει έννοια η αναφορά. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ή θεωρούν ορισμένοι ότι δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Και παρακαλώ θέλω μια σαφέστατη απάντηση. Ευχαριστώ κύριο Σεντακόφσκι. Ευχαριστώ. Γιατί πολύ καλά προφέρατε το όνομά μου. Είναι δύσκολο, το ξέρω, Σεσίλια. Θα μιλήσω γερμανικά. Καλύτερα. Δεν συμφωνώ και θέλω να επικρίνω το ότι δεν έχουμε πάρει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ισχύει αυτό που ο κύριο Ρόλ. Τους ρωτήσαμε κατά την ακρόαση δύο-τρεις φορές τι μπορούμε να κάνουμε. Στην Τσεχία ε, εδώ και δέκα χρόνια έχουμε λάβει πολλές αναφορές και ξέρουμε ότι είναι αρνητικό για την Ευρώπη να υπάρχει αυτή η αποφυγή ευθυνών. Αυτή η αλλαγή στην ώρα δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, στις μεταφορές προβλήματα και σύγχυση γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να μας δοθεί απάντηση. Υπάρχουν πολλές μελέτες που πιστοποιούν ότι κάνει ζημιά στην υγεία μας η αλλαγή ώρας. Πόσο θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη για να μας δοθεί απάντηση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να καταργήσουμε αυτήν την ε, θερινή ώρα. Έχουν υποβληθεί 11 αναφορές ήδη. Από την Τσεχία θα μπορούσα να σας στείλω και άλλες πολλές. και πολλές από αυτές ε, έχουν λάβει πολλές υπογραφές. Ορισμένες έχουν υπογραφεί από 100.000 άτομα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μας δοθεί απάντηση. Όπως είπε και ο Πάβελ Σβόμποντα, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, πάνω από 200 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κατά της θερινής ώρας. Άρα η πρωτοβουλία αυτή έχει όλο και ευρύτερη υποστήριξη. Επαναλαμβάνω ότι κάθε φορά όταν εφαρμόζεται κάθε χρόνο η αλλαγή ώρας λαμβάνουμε όλο και περισσότερες αναφορές. Σας ευχαριστώ πολύ που ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα. Και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη σωστή απάντηση. Να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κλίν έχει μάλλον ολοκληρωθεί ο κατάλογος ομιλητών. Ενδιαφέρον εδώ είναι ότι έχουμε τόσες πολλές αιτήσει και σχεδόν όλες είναι από τη Γερμανία. Γιατί? Πολίτες ανά την Ευρώπη ε, έχουν ευαισθησία σε αυτήν την αλλαγή ώρας, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μόνο από τη Γερμανία έρχονται οι αναφορέ, εκτό από μία-δύο εξαιρέσει. Είναι περίεργη αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί. σω είναι και πολύ σκληρό το λόμπι εδώ πέρα για του πολίτε. Δεν ξέρω. Γνωρίζω όμω ότι πολλέ φορέ έχει κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει απαντήσει και ακόμα δεν το έχει πράξει. Αυτή είναι η δική σας δουλειά. Παρακαλώ να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Και υπάρχει και το προφορικό ερώτημα που θα έρθει στην Ολομέλεια. Και αυτό σημαίνει, ή μάλλον εγώ προτείνω, να περιμένουμε την απάντηση στο προφορικό ερώτημα και ανάλογα με την απάντηση που θα λάβουμε, Μπορούμε εκείνη τη στιγμή να αποφασίσουμε να κλείσουμε τις αναφορές ή να τις διατηρήσουμε ανοιχτέ. Ανάλογα λοιπόν με την απάντηση που θα λάβουμε. Δεν βλέπω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, συμφωνούμε. Ωραία. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Α, προτιμάτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην απαντήσετε αυτή τη στιγμή. Μπορείτε απλώς να μεταφέρετε ε, το μήνυμα αυτό, ότι πραγματικά περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επόμενη αναφορά έχει αναβληθεί. Πάμε στο σημείο 11. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον. Να δώσουμε το λόγο απευθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κούντε Λάγκε. Ή Ιωάννα Βουλέσκου. Παρακαλώ. Κούντε Λάγκε. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής. Αυτή η αναφορά πράγματι αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο συγχρονοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και εδώ θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ουσιαστικά η αρχή διαχείρισης ορίζεται από το κράτος μέλος, αυτή που είναι υπεύθυνη μάλλον για τη διαχείριση των προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνη αυτή η αρχή για την επαλήθευση, επιτόπου επαλήθευση για τα προγράμματα. Δεν γίνεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Αρχή να μας, δώσει, να μας ενημερώσει για αυτό το project, επειδή την προηγούμενη φορά τότε εξέτασε η Επιτροπή, ακόμα δεν είχε οριστικοποιηθεί και κάποια ζητήματα έπρεπε να λυθούν από τον ανάδοχο και τον δικαιούχο. Σήμερα λάβαμε επιβεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι έχει ολοκληρωθεί, οριστικοποιηθεί το project. Η σύνοψη του προγράμματος αναφέρεται και στα παράπονα στις καταγγελίες του αναφέροντος, όμως επιβεβαιώνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ε, επιληθεί. Και σημαντικό επίσης είναι ότι λάβαμε δύο εκθέσεις για την υποδοχή έργων από την αρχή διαχείρισης. Η πρώτη από το 2012 ε, υποαίρεση υποδοχής έργων. Υπήρχε και ένας κατάλογος ε, των ολοκλήρωση έργων και ο ανάδεχος έλαβε προθεσμία τριών ετών ακόμα για να οριστικοποιήσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Και λάβαμε και αντίγραφο της τελικής υποδοχής του παραλαβής μάλλον του έργου από το 2015, πριν από ένα μήνα. Και εδώ καταλήγει η έκθεση ότι όλα οι εργασίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών. Επομένω, όλα τα ελαττώματα που είχαμε εντοπίσει στο παρελθόν έχουν όλα διορθωθεί. Ένα νέο στοιχείο που πρέπει να επισημάνω είναι την, την περασμένη Παρασκευή, αργά το απόγευμα, ο αναφέρον έστειλε και πάλι ε, mail ότι δεν υπήρξαν μέτρα για τη βελτίωση της ε, ποιότητας ή ότι ήταν σημασία σε αυτές οι βελτιώσεις. Δεν καταφέραμε να διασταυρώσουμε αυτές τις πληροφορίες ε, με την αρμόδια αρχή μέχρι σήμερα βεβαίως. Όπως και να έχει, η πρωτοβουλία της Επιτροπής εδώ δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από την αρμόδια αρχή να επαληθεύσει ότι έχει κλείσει και ολοκληρωθεί το έργο. Όπως και να έχει, η αρχή υλοποίηση η προθεσμία περίοδος υλοποίησης του προγράμματος 7-14 είναι μέχρι φέτος το Δεκέμβριο και η αρμόδια αρχή πρέπει να υποβάλει την τελευταία έκθεση για ολόκληρο το πρόγραμμα μέχρι το Μάρτιο 2017. Ένα έτος και τρεις μήνες μετά το πέρας για να μας ενημερώσει για όλα τα επιμέρους στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμεί Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Και τώρα πραγματικά χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να μου πείτε τι πρέπει να κάνω με αυτή την αναφορά. Ο κύριο Μαχτά. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε από μόνη τη. Υπάρχει ένα νέο στοιχείο στην όλη υπόθεση. Πρέπει να επαληθεύσουμε τι έχει πει αυτό ο αναφέρον πριν κλείσουμε την αναφορά. Αυτή είναι η δική μου πρόταση γιατί βλέπω άλλη λύση. Πίτερ, ζήτησε το λόγο. Έχω αμφιβολίες, καταλαβαίνω τον ε, αναφέροντα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχει έλεγχος κατά τη διάρκεια του έργου, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα, αν λείπει τώρα κάποιο τεχνικό στοιχείο για παράδειγμα, κάποιο κάλυμα, αλλά πρέπει να δούμε ποιος ελέγχει, ποιος ε, έχει την τεχνική ευθύνη, ποιος είναι ο επιβλέπων. Συνήθως λέμε ότι θα μπορούσαμε να την κλείσουμε αυτήν την αναφορά και ο, ο αναφέρον πρέπει να απευθυνθεί στις περιφερειακές αρχές. Τώρα αν δεν λειτουργεί κάτι, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να ψάξουμε μέχρι το τελευταίο σωλήνα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λειτουργούν σε άλλο επίπεδο αυτά. Στην ουσία εγώ θα ήθελα να μου πει, θα ήθελα να μου δώσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες, ε, ε, να μου δώσει λέω περισσότερες πληροφορίες ε, ο ετών ε, δηλαδή να μας δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία, πιο εμπεριστατωμένα. Ε, επομένως, ε, αν θέλετε να σας πω, ναι, εγώ θα ήθελα να παραμείνει για την ώρα ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ωραία. Έχει ολοκληρωθεί μάλλον ο καταλόγος ομιλητών. προς τη Γραμματεία. Ο αναφέρον μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας από το 2011 και το έστειλε αυτό μόλις χθες. Χθες. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να δούμε κατά πόσο όλα αυτά τα στοιχεία ισχύουν, αν οι φωτογραφίες είναι από εκεί ή από κάπου αλλού. Όλα είναι δυνατά. Μπορούμε λοιπόν να στείλουμε πίσω το παλάκι στην Επιτροπή και να μας ενημερώσει όταν ε, έχει νέα στοιχεία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, κάτι ακόμα θα ήθελα να αναφέρω. Υπήρξαν και επιτόπιες επισκέψεις από την αρμόδια αρχή και από, τις, ε, από την κρατική υπηρεσία για το δικό δίκτυο. Νομίζω το 2012 έγινε αυτό και υπήρξαν μόνο μικρές ε, αδυναμίες ε, του έργου, που από ό,τι ξέρουμε τώρα έχουν διορθωθεί. Αυτό προκύπτει την τελική έκθεση. Αν το θέλετε, βεβαίως μπορούμε να στείλουμε επιστολή στην αρμόδια αρχή για να δούμε αν το έχει επαληθεύσει ή αν μπορεί να υπάρξει εκ των υστέρων ε, του έργου. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, τα γενικά ζητήματα έχουν λυθεί. Ίσως όμως υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες και αυτές τις λεπτομέρειες να μας στέλνει. Ίσως. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση της Ελεονόρ να μην ανοιχτεί η αναφορά και η πρόταση του Πίτερ να την κλείσουμε. Τι θέλετε να κάνουμε. Όχι, όχι. Όχι, συμφωνώ με την Ελεονόρα. Καλή πρότασή της. Η πρότασή μου είναι ότι όταν θα έχουμε την πληροφόρηση αν μας πει η γραμματεία ότι όλα επαρκούν, τότε θα μπορούσαμε να το κλείσουμε μέσω διαδικασία σημείου Β. Εάν θεωρήσουμε ότι είναι, επαρκής, ότι η πληροφόρηση και ότι όλα είναι εντάξει, να αφήσουμε λοιπόν τώρα ανοιχτή την αναφορά και να αφήσουμε τη γραμματεία να μας κάνει πρόταση για το πώς θα αποφασίσουμε με βάση την πληροφόρηση που θα λάβει. Ωραία, θα κάνουμε ακριβώς αυτό που πρότεινε ο Πίτερ. Η γραμματεία θα εξετάσει τις λεπτομέρειες και μετά θα δούμε αν θα κλείσουμε την αναφορά ή θα ερευνήσουμε περαιτέρω στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής. Ωραία, συνάδελφοι, κλείνουμε εδώ. Καλή όρεξη και σας περιμένω αναζωογονημένους το απόγευμα.